δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στον εισηγητή, τον κύριο Σόποδα, για τέσσερα λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σας πληροφορήσω για το περιεχόμενο της έκθεσης Επιτροπής Νοεμικών Θεμάτων για την προστασία των δικαιωμάτων ε, διανοητική ιδιοκτησία, το σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω έχω τονίσει και στο παρελθόν, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που η Επιτροπή Γιούρι Νομικών Θεμάτων ω σύνολο δέχτηκε την προσέγγιση μου για το ζήτημα αυτό, που συνίσταται στο να εστιάσουμε για την έκθεση για το σχέδιο δράση και όχι να συζητήσουμε άλλα άσχετα θέματα. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει γενική συμφωνία στο ότι η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας είναι θετική για την πολιτιστική πολυμορφία αλλά και για τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό εμείς χαιρετίζουμε τις κινήσεις που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βελτιώσει την κατάσταση αυτή. Επίσης χαιρετίζουμε την προσπάθεια της Κομισιόν να παρουσιάσει τα εργαλεία τα οποία θα βασίζονται σε μια καλύτερη κατανόηση του πώς λειτουργεί το σύστημα αυτό και τα οποία θα δημιουργήσουν μια βελτιωμένη διαδικασία διαβούλευσης με τους εμπλεκομένους. Νομίζω ότι η γενική συνένεση και η γενική κατανόηση όλων αυτών των πλευρών θα μας, θα μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε ένα πραγματικά αποτελεσματικό σύστημα για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την εφαρμογή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι μια η πληροφοριακή εκστρατεία έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει μέσα στην στατική αυτή του σχεδίου δράσης. Θα πρέπει επιπλέον να συμφωνήσουμε τα βασικά δικαιώματα <clears throat> και προφανώς ξέρω ότι η κυρία Πίτροπος σέβεται όλα αυτά τα δικαιώματα αλλά αυτό το οποίο μας ε, ενδιαφέρει είναι η γενικότερη αποδοχή από το ευρύ κοινό και στον τομέα λοιπόν των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο ζήτημα αυτό. Θέλω να υποστηρίξω επίσης και την αντιμετώπιση της Επιτροπής. Πιστεύω ότι υπάρχει μια συνένεση στο ότι εάν θέλουμε να βοηθήσουμε οι οποίοι πρέπει να αγωνιστούν εναντίον της παραβίασης των πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει να είμαστε πιο ενεργοί στα θέματα αυτά. Και εγώ προσωπικά θέλω να υποστηρίξω την προσπάθεια της Κομισιόν να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν νομίζω <clears throat> ότι αυτό είναι μια ε, προνομιακή μεταχείριση. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα από τα πολλά ε, εγχειρήματα σε ένα μεγάλο χώρο που, όπου θα πρέπει εμεί να βελτιώσουμε την κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα λοιπόν εφαρμογής των διανοητικών δικαιωμάτων Δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία είναι πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζω ότι και η Κομισιόν θα συμβάλλει σε αυτό το εγχείρημα με ουσιαστικό τρόπο. Η εφαρμογή του σχεδίου δράση θα πρέπει να επιταχυνθεί, θα πρέπει να έχει την απαραίτητη ευκαμψία ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει και τι νέε εξελίξει και θα πρέπει να βασίζεται σε δικαιολογημένες ενέργειες που θα οδηγήσουν σε μια καλύτερη προστασία για τους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτή είναι και η βάση και ο ακρογωνιαίος λίθος όλης της στρατηγικής μας, να ενισχύσουμε την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Ελπίζουμε από τον Ιούλιο του 2016 η Κομισιόν θα βέλθει ενώπιόν μας να μας δώσει τα πρώτα αποτελέσματα αυτού του σχεδίου δράσης. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε τώρα με τη δικασία Catch the Eye. Ο κύριος Μαριάς έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας αποτελεί κινητήρια δύναμη για την απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα έχει ζωτική σημασία για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας πρέπει να συμπεριλάβει την υιοθέτηση μιας προσέγγισης που συνίσταται στην παρακολούθηση της γραμμής του χρήματος προκειμένου να χτυπηθούν οι παραβάτες των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που διακινούν παραποιημένα πειρατικά προϊόντα μέσω του διαδικτύου. αυτό είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις εθνικές οικονομίες. από την άλλη πλευρά πρέπει να υπάρξει μια δίκαιη ισορροπία συμφερόντων μεταξύ των κατόχων των δικαιωμάτων αυτών και των τελικών χρηστών. τέλος σε μια φάση οικονομικής κρίσης που πλήττεται η χρηματοδότηση του πολιτισμού λόγω περικοπών που επιβάλλει η μερκελική δημοσιονομική προσαρμογή θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη στήριξη του πολιτισμού από την πλευρά της ευρωπαϊκής ένωσης. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να τονίσω δύο σημεία. Πρώτον, η δημιουργικότητα και η καινοτομία αποτελούν εγγύηση για μια ποιοτική οικονομική ανάπτυξη και εγγυώνται κατά αυτόν τον τρόπο το μέλλον μας. Χωρίς δημιουργικότητα, χωρίς έρευνα δεν μπορούμε να έχουμε οικονομική ανάπτυξη. Η δημιουργικότητα, η έρευνα και η κοινοτομία όμως απαιτούν και μία προστασία των δικαιωμάτων διονυτικής ιδιοκτησίας. Από την άλλη, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν πραγματικά τη ραχοκοκαλιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν συνδυάσουμε λοιπόν τις δύο αυτές σκέψεις, τότε πραγματικά θέλουμε να έχουμε μία δημιουργικότητα, η οποία όμως να περνάει κυρίως και μέσα από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και το σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει να κάνει με την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων διοντικής διοκτησίας θα πρέπει ακριβώς να προστατεύει και τη δημιουργικότητα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι πολύ σημαντικό να καλύψουμε και να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησία. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι έχει να κάνει με τα συμφέροντα των καλλιτεχνικών δημιουργών και όχι με το, τα συμφέροντα των ε, ενδιάμεσων επιχειρήσεων που θεωρούν ότι η καλλιτεχνική δημιουργία είναι απλώς ένα εμπόρευμα το οποίο θα πρέπει <clears throat> να εκμεταλλεύονται με οικονομικούς όρους γνωρίζοντας την αξία των πολιτιστικών προϊόντων, όλοι αυτοί οι οποίοι είναι καλλιτεχνικοί δημιουργοί θα πρέπει να έχουν μια αξιοπρεπή προστασία σε επαγγελματικό επίπεδο. Δεν πρέπει απλώς να έχουν μια θέση εργασίας. Πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν με ευφύ τρόπο <clears throat> αυτή την προστασία. Και εξάλλου όλα τα άτομα θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να απολαμβάνουν τα πολιτιστικά προϊόντα, να έχουν πρόσβαση στη γνώση και φυσικά με την προϋπόθεση ότι θα δίνουν μια αντίστοιχη αμοιβή στους καλλιτεχνικούς δημιουργούς χωρίς όμως να την κατατρών η ενδιάμεση. Ευχαριστώ πολύ. Άρνοτ, κύριε Πρόεδρε. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου πέντε βουλευτές ή μόνο πέντε βουλευτές από τους 751 για τη δεύτερη συζήτηση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Εγώ θέλω να προχωρήσω αυτό που είπα προηγουμένως, ότι πρέπει να ενισχύσουμε τα συμφέροντα των μικρών επιχειρήσεων. Οι Βρυξέλλε έχουν πιο πολλούς λομπίστε από ότι η Washington στις ΗΠΑ. Πάνω από 30.000 λομπίστε. 40 για κάθε ευρωβουλευτή λοιπόν. Γι' αυτό οι εκλογέ μου διαμαρτύρονται για την πίεση των μεγάλων επιχειρήσεων για θέματα όπως το TTIP. Και έχουν δίκιο που το κάνουν. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή λοιπόν για το γεγονό ότι υποστήριξε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, ιδίω στου τομεί όπω η ανάπτυξη λογισμικού. Οι μικρέ επιχειρήσει μπορεί να συνθλιβούν από τι νομικέ υπηρεσίε των μεγάλων επιχειρήσεων. Εγώ <clears throat> δεν θέλω να με πιέζουν οι μεγάλε εταιρείε, αλλά οι εκλογή μου και μόνο. Ευχαριστώ, λέω Η Επίτροπος τώρα έχει το λόγο. Πρόεδρε, αξιότιμοι προβουλευτέ, σας ευχαριστώ πολύ για τις παρεμβάσεις σας και για τη δουλειά που έχετε κάνει για την έκθεση αυτή και ιδιαίτερα τον κύριο Σφόποντα. Έχει συνεισφέρει πολύ σημαντικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή την κοινή προσπάθεια για την πρόθεση της καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την δράση της στην καινοτομία όσον αφορά το νομοθετικό πλαίσιο σε το τομεί κλειδί για την διανοητική ιδιοκτησία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε στοχευμένε δράσεις για να ενισχύσει τα δικαιώματα αυτά και στην εσωτερική αγορά. Αντιμετωπίζουμε μια δύσκολη και περίπλοκη πραγματικότητα οι εμπορικές δραστηριότητες μερικές φορές δυσχεραίνονται και γι' αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως από άτομα αλλά και από επιχειρήσεις που κανονικά πρέπει να αποφελούνται από τα δικαιώματα αυτά και να μην αποτελούν εμπόδιο. Η εμπορική διάσταση λοιπόν και η σχέση της με την παρεπόδεση της διονυτικής ιδιοκτησίας απαιτεί δημιουργικότητα, απαιτεί καινοτομία και εφευρετικότητα. Πρόκειται για θεμητές δουλειές που πολλές φορές χάνονται, χάνεται κέρδος. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να εφαρμόσουμε κατάλληλα μέτρα κατά τέτοιων δραστηριοτήτων σε βάρος της διοντικής ιδιοκτησίας. Τα μέτρα που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον Ιούλιο του 2014 συμπεριλαμβάνει μη νομοθετικά μέτρα. Κάποια από αυτά προωθούν την ε, ασφάλεια, την καινοτομία και την ε, δημιουργικότητα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Όπως φαίνεται και από την έκθεση του κύριου Σβόποτα, οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της επιβολής των δικαιωμάτων διονοητικής ιδιοκτησίας πρέπει να συνεχιστεί και κυρίως στα εξή σημεία. Προστασία των καταναλωτών ε, κατά ε, προστασία μάλλον από παραπημένα προϊόντα. Ε, βοήθεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να δούμε ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος των μεσαζόντων. Ε, εφαρμογή της, ε, της επιμέλειας. Υπό τους επιτρόπους λοιπόν τους αρμόδους για τα θέματα αυτά παρακολουθούμε τη... τις εργασίες σας όπως επίσης και το τι κάνει ο κλάδος για όλους αυτούς τους τομείς. Η στήριξη του σώματός σας είναι ζωτική σημασία καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Θέλω όμως να πιστήσω την προσοχή σας και στο γεγονός ότι παρά την καλή πίστη πολλών πρωτοβουλειών και του προγράμματος δράσης του 2014 η εφαρμογή των ε, δικαιωμάτων αυτών μπορεί να απαιτεί και νομοθετικές αλλαγές. Έχουμε τη στρατηγική για την ψηφιακή αγορά και περιλαμβάνεται και η πνευματική ιδιοκτησία. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι άλλου είδους δικαιώματα δυνατικής ιδιοκτησίας έχουν μικρότερη σημασία γιατί αλλιώς αυτό θα ήταν σε βάρος τη ευρωπαϊκή οικονομίας. Συνεπώς, σε επόμενους μήνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προχωρήσει σε αξιολόγηση της συνολική λειτουργίας ε, της ε, επιβολής των δικαιωμάτων δυνατική ιδιοκτησία. Αν διαπιστώσουμε ότι χρειάζονται αλλαγές, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επικεντρωθεί ακριβώς σε αυτό στο μέλλον. Εν κατακλείδη, θέλω να ευχαριστήσω και πάλι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το γεγονός ότι θετικά αντιμετώπισε το πρόγραμμα δράσης και ελπίζω να το εγκρίνετε αύριο. Ελπίζω πραγματικά ότι η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα των δικαιωμάτων κοινωτικής ιδιοκτησία και επιβολής τους θα συνεχιστεί προς όφελος της καινοτομίας, της δημιουργικότητας, της απασχόλησης υπέρ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστούμε πολύ την Επίτροπο. Ε, ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Θα ψηφίσουμε